Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εκ μέρους των Πρασίνων και στην έκθεσή σας, ιδίως στο σημείο και στο εδάφιο που αναφέρεστε στο άρθρο 2 της συνθήκης, και τονίζει το σεβασμό των δημοκρατικών αξιών, δείτε εδώ υπονομεύονται, και την διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση όντως. Αλλά στην ομάδα των Πρασίνων, όπως και εσείς, ε, θα φροντίσουμε να ενισχύσουμε την έκφραση εδώ, διότι γι' αυτό ακριβώς θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Θέλουμε να ενισχυθεί η μία στο κάτω δικαίου με κάποιες τροπολογίες, τροπολογίες οι οποίες ε, θα κάνουν πιο ανάγλυφη τη θέση σας και μια δεδομένη, μια βασική τεκμηριωσή για όλες τις ε, υποθέσεις διαφθοράς που έχουν εντοπιστεί. Η συστημική διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Να περιμένετε λοιπόν μια σωρία από τροπολογίες από πλευράς μας επίσης. Θα υποβάλουμε κάποιες ακόμη πιο γενικόλογες τροπολογίες, οι οποίες καταρτίζουν ε, ένα σχετισμό μεταξύ της έλλειψης διαφάνειας ό,τι αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κοντιλίων, και την, ε, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κακοδιαχείριση στα συμφέροντα της κοινωνίας. Μιλήσαμε στην ε, κεκλεισμένο των θυρών ε, συνεδρίαση για τους διαγωνισμούς με έναν μόνο προσφέροντα. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που πρέπει να το σχολιάσουμε στην εκθεσή μας και να συμπεριληφθεί. Πρέπει να δοθεί κατάλληλη έμφαση. Επίσης θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για τον τρόπο που οι θεσμοί στην Ουγγαρία δεν λειτουργούν σωστά σε ό,τι αφορά τον, ε, την εφαρμογή της νομοθεσίας και τις ε, διαδικασίες ελέγχου. Ο δημόσιος εισαγγελέα ε, και η δικαστική αρχή δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Οι έρευνες της Όλαφ ή των ερευνητών δημοσιογράφων ε, καταδεικνύουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να επικρίνουμε την ε, αποτυχία των ουγγρικών ε, θεσμών στο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την εκθεσή σας. Νομίζω είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ κύριος Ιβάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πήγαμε μαζί σε αυτήν την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στην Ουγγαρία και θέλω να προσθέσω ότι είναι σημαντικό να προστατευθούν οι σε ερευνητές δημοσιογράφοι και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μέχρι τώρα δεν τους έχει επιτραπεί να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που καταφέρουν να εξεύρουν για επιχειρηματίες και για μεγάλα συμφέροντα στη χώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Στην Ουγγαρία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κόσμος που έχει δικαίωμα να είναι δικαιούχος σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορεί όμως ένα κράτος μέλος να μην ε, τηρεί τις υποχρεώσεις του. Θα πρέπει λοιπόν η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθείται και από κάποιε ε, υποχρεώσεις. Διαφάνεια ω προς το πού πηγαίνουν τα κονδύλια, πώ εκτελούνται, τι επιδόσεις υπάρχουν, διότι είδαμε ότι 60% των επενδύσεων έχουν ε, βασίζονται σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό δεν ταιριάζει με τις αντιευρωπαϊκές τοποθετήσεις τη κυβέρνηση στην προεκλογική τη εκστρατεία και γενικότερα. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν ε, αναφέρονται στις προεκλογικέ εκστρατείε. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται λοιπόν για τέτοιους σκοπούς. Και δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για αυτό το κράτος μέλο, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και λίγα λόγια για το θέμα της διαφθοράς στην ε, χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εγώ παροτρύνω την Όλαφ να διεξεγάγει ακόμη περισσότερες έρευνες για να δει πού κατέληξαν τα κονδύλια και πόσο σημαντικό είναι το φαινόμενο της διαφθοράς. Εάν τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι αντικείμενο κακοδιαχείρισης και δεν ε, υλοποιούνται τα ευρωπαϊκά έργα, εάν ο κόσμος που... Ε, οι θύνοντες της κυβέρνησης απλώς ε, βάζουν στην τσέπη αυτά τα χρήματα, αυτό είναι κάτι που θα βλάψει το ίδιο το κράτος ε, εντός του οποίου συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν θα ανακάμψει. Και υπάρχει και δυσμενής ε, εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσμενής επιπτώσεις για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είναι λογικό τα ευρωσκεπτιστικά τα ευρωπαϊκά, τα αντιευρωπαϊκά κινήματα να κερδίζουν έδαφος. Αντί λοιπόν να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ουσιαστικά παρεμποδίζεται η θετική ανάπτυξη, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια για τη χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα... Άκουγα τη μετάφραση, με συγχωρείτε. Νομίζω το κείμενό σας είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Διότι χρειάζεται καλή διακυβέρνηση για να καταπολεμηθεί η κακοδιαχείριση κοντελίων. Στην ε, Ουγγαρία υπάρχουν πολλέ αμφιβολίε για το πόσο αυτό ισχύει. Και γι' αυτό θα επικρίνουμε κιόλα. Στην πρώτη παραγραφή τη εκθεσή σα, όπου αναφέρεστε σε αυτό, θα μπορούσατε να είστε ακόμη πιο δρυμία. Και γι' αυτό θα υποβάλουμε σχετικά τροπολογίε. Έπειτα χρειάζεται και πρόληψη πέρα από την ε, καλή διακυβέρνηση. Πρέπει να δοθεί περιθώριο στους καταγγέλλοντες και τους ερευνητές δημοσιογράφους να δράσουν. Κάτι θα πρέπει λοιπόν να υποθεί πιο ρητός και γι' αυτό. Και το τρίτο που χρειάζεται είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το ίδιο το γεγονός που το δηλώνετε και στην έκθεσή σας, ο 36% των ε, διαγωνισμών είναι διαγωνισμοί με έναν προσφέροντα, με μία μόνο προσφορά για την ανάθεση του έργου, είναι μια καθοριστική πληροφορία. Πρέπει να επιληφθεί όλα. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να γίνουν σχετικέ συστάσει και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ε, έκθεσή μα, αλλά βρίσκω το κείμενο μια πολύ καλή βάση και ανεπομονώ να διαβάσω τι τροπολογίε των πρασίνων όπω μα προαναγγέλθηκε. Ελπίζω να μπορούμε να τι στηρίξουμε όλε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε από τους συναδέλφους παρατηρήσεις, πολιτικά επιχειρήματα, κυρίως μας προειδοποίησε η Πρόεδρος ότι δεν θα πρέπει να προβάλλουμε πολιτικά επιχειρήματα. Δεν ξέρω αν είναι προνόμιο μόνο στην Επιτροπή αυτή των Πρασίνων της Αριστεράς. Δυστυχώς το κείμενο που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι σχέδιο γνωμοδότησης, είναι μάλλον σαν ε, ε, μία σειρά παρατηρήσεων χωρίς να υπάρχουν σοβαρά ίσως επιχειρήματα. Υπάρχουν Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις για το σύνταγμα στην Ουγγαρία από κάποιο δανό, ο ε, κάτι έλεγε για το... κάποια δανή, η οποία κάτι έλεγε για το πρώτο άρθρο του συντάγματος. Βεβαίω είχε κάνει λάθο, γιατί μινούσε για τον πρώτο στίχο του εθνικού ύμνου τη Ουγγαρία και όχι για τον πρώτο άρθρο του συντάγματο nem Υπάρχει λοιπόν πραγματικά κάποια λανθασμένη άποψη. Είπατε ότι όταν έχουμε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο στις κρατικές προμήθειες, αναρχόμαστε σε ποσοστό γύρω στο 36%. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτή όλη αυτή η οι διαγωνισμοί, όλες αυτές οι αναγγελίες προσφορών. Είναι σε γνώση όλου του κόσμου. Έχει πέσει το ποσοστό από το 36% 24%. Δεν νομίζω ότι πολλές άλλες χώρες μπορούν ε, να μιλήσουν για, τέτοιου είδους, για, τέτοιο, για τόσο χαμηλά ποσοστά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνονται τέτοιου είδους λάθη σημαντικά. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Ουγγαρία, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επίσημη αξιολόγηση γίνεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 15 χρόνια, λαμβάνεται υπόψη και διαπιστώνουμε ότι βελτιώνονται κάθε χρόνο τα ποσοστά και οι αριθμοί που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων. Ακόμη και τα πρώτα χρόνια της ε, ε, προσχώρησης είχαμε υψηλά ποσοστά διαφοράς, αλλά μειώθηκαν τα ποσοστά. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σχεδόν αστείο αυτό που λέγεται για αυτά τα κέντρα διαφθοράς που το έχουν οι ακτιβιστές πολιτικοί. Επαγγελματίες δηλαδή. Τι εννοούμε. Αυτή η οργάνωση, στην οποία αναφέρεται, κάνει πολιτικές δηλώσεις ανακοινοθέντα τον τύπο, αλλά δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας στην ε, Ουγγαρία που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτά τα οποία λέει αυτή η οργάνωση. προσπαθούν να περιγράψουν την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για κάποια θέματα. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν κανένα σχετικό έγγραφο στη διάθεσή τους που να αποδεικνύει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στα προγράμματα τα οποία, ε, τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να αποδείξουν κάτι τέτοιο ούτε να κάνουν συγκρίσεις. Βεβαίως, σε, υπάρχει υπερτιμολόγηση σε πολλές ε, περιπτώσεις, σε πολλούς ε, τομείς, σε πολλές χώρες. Όταν έχουμε να κάνουμε με συγκρίσιμες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται χρησιμοποιώντας παρεμφερή τεχνολογία. Αυτό το βρίσκεται σε όλες τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Ναι, Και πολλές φορές ε, ε, αυτά τα πράγματα πρέπει κανείς να μπορεί να τα αποδείξει. Στην Ουγγαρία, όσον αφορά τις κρατικές προμήθειε δημόσιες προμήθειες, είτε συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε χρηματοδοτούνται, είτε χρηματοδοτούνται από την αγορά, δεν είναι ανώτερες οι τιμέ. Επίσης, τελικά συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω ότι η, η Επιτροπή μας σκέπτεται να θεσπίσει αυστηρότητα, αυστηρότερα μέτρα έναντι κάποιας χώρας. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ μπορεί να ισχύσει και η αρχή του opt-out. Τώρα τι να πω, ότι παντού υπάρχει διαφθορά σε όλες τις χώρες. υπάρχουν και κάποιες ε, βόρειες χώρες, τις οποίες δεν μπορεί κανείς να πει ότι θεωρούνται χώρες τις οποίες υπάρχει διαφορά. Είναι λοιπόν απαράδεκτο. Με έναν θεσμικό όργανο που βασίζεται στην ε, ε, εθελούσια συνεργασία, την ενισχυμένη ε, συνεργασία, να κάνει τέτοιου είδους παρατηρήσεις και καταγγελίες. Ε, nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης δεν θα είναι στην ε, ίδια του μορφή στη συνέχεια γιατί θα συμπεριληφθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με το θέμα και βέβαια θα κατατεθούν σχετικές τροπολογίες. Η Ουγγρική κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, θέλει να οροποιήσει κάποια στατιστικά στοιχεία. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά πώς έχει αυτή η κατάσταση με τους ε, μοναδικούς ε, ε, υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι τελικά παίρνουν τις συμβάσεις αφού έχουν αποκλειστεί με διάφορους τρόπους και μέσα οι υπόλοιποι υποψήφοι. Και πρόκειται για εταιρείε που είναι πολύ κοντά στην πολιτική ελίτ αυτοί που παίρνουν, αυτές που παίρνουν τις προσφορές και τις συμβάσεις. Υπάρχουν ΜΚΟ που δέχονται ιστερική ε, κριτική γιατί παρουσιάζουν κάποια στοιχεία για την ε, ε, κυβέρνηση που θέλει να τα κρύψει. Σε ό,τι αφορά την υπερτιμολόγηση. Τα ογκρικά επενδυτικά έργα είναι πολύπλοκα. Επίτηδες δε είναι τόσο πολύπλοκα ακριβώ για να μην υπάρχει περίπτωση συγκρισιμότητας. Γι' αυτό η έλεγχη πρέπει να είναι σε μεγάλο βάθος για να εντοπίσουν τις υπερτιμολογίες αυτές. Όμως κάποιες από τις τιμές των προσφορών είναι πραγματικά αστρονομικές. Σε ό,τι δεν αφορά τη γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Νομίζω ότι μία μια κυβέρνηση δεν θα μιλήσει για θέμα εθνικής κυριαρχίας. αλλά παίρνουν δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοοικονομικής υποστήριξης, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις υποψίες. Οπότε φαντάζομαι ότι θα προσχωρήσουν με τα χαράς στο γραφείο εισαγγελία. Οι χώρες όμως που δεν θα προσχωρήσουν δεν ωφελούνται από ό,τι φαίνεται από τον νοσιακό προπολογισμό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε όμως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έλεγχου. Η κυρία Ρενκό από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Τζάστ. Thank you, Madam Chair, uh, for giving us the floor. Good morning, everybody. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ως προς τα όσα ακούσαμε από τις διάφορες ε, παρεμβάσεις, απλώς να επαναλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαφυλάξει τι ευρωπαϊκέ αξίε και το ευρωπαϊκό δίκαιο και βεβαίω όσα προβλέπει η Χάρτα των Θεμελιωδιών Δικαιωμάτων. Γι' αυτό χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την διαφθορά στα κρατημέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βάσει της ε, έκθεσης αναχώρα μπορεί να εκδώσουμε συγκεκριμένε αναχώρα σύσταση ε, για τα ενδιαφερόμενα κρατημέλη και πολύ πρόσφατα στις 7 Μαρτίου φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις φετινές αναχώρα εκθέσεις όπου ανέλησε τις βασικές προκλήσεις ό,τι αφορά τη διαφθορά για διάφορα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανόμενες της Ουγγαρίας. Στην έκθεση αυτή Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε αναφορές για τους ε, ιδιαίτερους κινδύνους και τα κενά που έχουν εμποδίσει τις επενδύσεις, την σωστή απόδοση των πόρων, τις οικονομικές ε, καλές επιδόσεις και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ των Ελευθεριών του Πολίτη με την ενδεχόμενη σύνταξη βάσει του άρθρου 7.1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω από πλευρά μου αυτά είναι όσα είχα να πω. Ας ακούσουμε και την Όλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά της Όλαφ, απλώς να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται κάποια διορθώση δεδομένων ε, στα στοιχεία που μεταδώσαμε στη γραμματεία για τη σύνταξη της έκθεσης, μερικές μικρές διορθώσεις για το 2016. όπου θα αναλυθεί δράση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εθνικό επίπεδο για τις συστάσεις που αφορούν το δικαστικό κλάδο. Τα δεδομένα για το 2017 εξετάζονται τώρα. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να τα αποκαλύψω. Χρειάζεται έγκριση του Γενικού μας Διευθυντή, αλλά θα σας τα διαβιβάσουμε, Πρόεδρε, μόλις τα ετοιμάσουμε. Πέραν αυτών, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Και αν έχετε συγκεκριμένε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 5 Απριλίου, το επαναλαμβάνω. Φαντάζομαι ότι θα λάβω πολλές ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Έχουμε το επόμενο σημείο παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Καμαδελταρή και πότε θα έρθει. Στις 11 έπρεπε να είναι εδώ, απαντάει κάποιος από την Κομισιόν. Ναι, γι' αυτό ρωτάω, λέει η Πρόεδρος, ε, ισχύει αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, 12, ε, σημείο 12 σημερισιάς διάταξης. Ανταλλαγή απόψε λοιπόν με το Γενικό Διευθυντή της Χαμαδέλτα Ρέγκιο σε σχέση με την πολιτική συνοχή πάλι για την Ουγγαρία-Πολωνία και συν Σλοβακία-Τσεχική Δημοκρατία από την προσχώρησή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την 7η έκθεση για τη συνοχή και θεωρήσαμε σημαντικό να συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο στη διάταξη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, έχουμε μια ώρα στη διάθεσή μας. Μπορεί κανείς να ψάξει να βρει το Γενικό Διευθυντή. já bych chtěl mluvit k tomu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 Καλημέρα συνάδελφοι. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε για την πολιτική συνοχή σε τρεις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για αυτές τις χώρες, τις τέσσερις. Από όσων ξέρω, 13 χώρες προσχώρησαν στην τελευταία διεύρυνση θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε όλες αυτές τις χώρες ή σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν τα κονδύλια στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Όταν μιλούμε για το ποσοστό απορρόφησης, γιατί πρέπει να εστιαστούμε μόνο σε αυτές τις τέσσερις χώρες ή γιατί κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών που εντάχθηκαν μετά το 2004 και τις προ... αυτές που εντάχθηκαν προηγούμενα. Στην ε, Τσεχία έχουμε λάβει μέχρι τώρα 24 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια δις από την ε, χώρα έχουμε κάποια προβλήματα απορρόφησης και δεν μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα, αλλά η κατάσταση όλο και βελτιώνεται και τα αποτελέσματα τώρα είναι καλύτερα και τα επιχειρησιακά προβλήματα, προγράμματα συγγνώμη, ίσως γίνουν προβληματικά. Το 2015 υπήρχαν προγράμματα ύψους 36 δις, κάποια από τα οποία συγχρηματοδοτούνταν και είμαστε από τις χώρες όπως και η Σλοβονία, η Πολωνία και η Ουγγαρία που αναπτυσσόμεθα με τους υψηλότερους ρυθμούς. Πολλές φορές έχουμε κατά 50% ποσοστά υψηλότερα όσον αφορά τη συνοχή απόψη άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, αλλά Όλε οι χώρε που χρησιμοποιούν τα κονδύλια συνοχή βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, παρά το γεγονό ότι υπάρχει οικονομική ύφεση. Επίση, θα ήθελα να αναφέρω ότι χθε είδαμε την έκθεση τη Επιτροπή τα της τη και Μόνο λίγες χώρες έχουν ε, υιοθετήσει μια σχετική στρατηγική, αλλά η Σλοβακία και η Ουγγαρία ήταν μεταξύ αυτών που υιοθέτησαν μια στρατηγική. Και βεβαίως με την αρεσιμότητα επίσης δεν είχαμε πρόβλημα για να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι τέτοιου είδους κονδυλίων. Και ένας από τους όρους, μία από τις προϋποθέσεις ήταν αυτό που αφορά τις ε, ε προσφορές, τις δημόσιες συμβάσεις. είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να μπορεί να προστατευτεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου προβλήματα. Αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς είναι να υπάρχει συνεργασία και καλύτερη σε προϋποθέσεις και οι χώρες μας προσπαθούν να είναι πάρα πολύ διαφανείς όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν. Ευχαριστώ. Μα δεν έχει υποστήριξει κανείς το αντίθετο μέχρι στιγμής. Απλά υπάρχει πρόβλημα σε κάποια ε, χώρες, μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες. Γι' αυτό και συζητούμε σήμερα για τέσσερα μόνα. Καρατέσουμε, δεν θα μιλήσουμε για τα επόμενα κάποια στιγμή. Ήρθε ο κύριος Μαρκ παρακαλώ. Κύριε Γενική Διευθυντά, έχετε το λόγο. Äh, äh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να μιλήσω. Είναι πράγματι κατάλληλη στιγμή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να πάρουμε απόσταση και να δούμε τη γενική εξέλιξη σε αυτά τα σημαντικά κράτη-μέλη και για, τη, για τους δικαιούχους, τους βασικούς δικαιούχους ε, της πολιτικής συνοχής από την προσχώρησή τους το 2004. Μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τα βασικά στοιχεία. Οι αλλαγές στο ΑΕΠ της Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διατεκομένη γραμμή. Αρχίζουμε από το σημείο 100 το 2014 και βλέπετε ότι η διατεκομένη γραμμή τελικώς είναι η πιο ε, επίπεδη ε, ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξελιχθεί λιγότερο θετικά από ότι το ΑΕΠ των χωρών αυτών. Βεβαίω πέραν αυτού βλέπετε και αρκετά σοβαρέ διαφορέ μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών. Η Ουγγαρία είναι πολύ κοντά στο μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι Η δημοκρατία της Τσεχίας είναι κάπως παραπάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο, είναι οικονομικά δυναμική και επίσης οι δύο πρώτοι, η Σλοβακία και η Πολωνία, είναι πάλι στήθος με στήθος στη διαφορά. Στην Πολωνία αυτό που ακόμη παραμένει αξιοσημείωτο είναι ότι η Πολωνία κατάφερε να περάσει από την οικονομική κρίση χωρίς καμία αρνητική, κανένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή μέχρι και το 2009 και 2010 είχαν ανάπτυξη, θα έλεγα βεβαίω, κατά τη δική μου άποψη, και χάρη στη σημαντική συμβολή ακριβώς σε εκείνα, τα χρονικά σημεία, χάρη λοιπόν στην ε, σοβαρή συμβολή της χρηματοδότησης ε, από το τέλος της περίοδου 2004-2006 και την αρχή της χρηματοδότησης από το 2007-2013. Εάν δείτε του συμπιλημένου αριθμούς της ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 έχει αυξηθεί κατά ένα 2,1%. Η Ουγγαρία δεν τα έχει πάει πολύ καλύτερα. 16% βλέπετε και η Πολωνία και η Σλοβακία είναι ε, πρωταγωνιστές, πρωταθλητές εδώ, φτάνουν περίπου το 60% της ανάπτυξης. Αυτά τα 13 χρόνια. Και βλέπετε ότι και οι πιο πρόσφατες τάσεις παρουσιάζουν ε, τις ίδιες, ε, τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ουγγαρία να είναι κάπως πιο κάτω από τα υπόλοιπα τρία κράτη-μέλη. Επόμενη διαφάνεια. Πώς έχουν μεταφραστεί οι αλλαγές αυτές σε αν, ε, κατακεφαλή ΑΕΠ και σε στοιχεία αγοραστικής δύναμης ό,τι αφορά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπει κανείς να έχει επιταχύνει και να προλαβαίνει το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Πολωνία και η Σλοβακία κάποια προσπάθεια από ήδη υψηλό επίπεδο διαβίωσης έχει πετύχει και η Δημοκρατία της Τσεχίας και πιο ταπεινά ξεκινώντας ως δεύτερη πιο ανεπτυγμένη μεταξύ των χωρών Βίζεγκραντ η Ουγγαρία, τελικά 13 χρόνια μετά, με σχετικούς όρους, γίνεται η λιγότερο ευημερούσα από τους τέσσερις. Η Πολωνία έχει προλάβει και έχει ξεπεράσει την Ουγγαρία. Οι αλλαγές σε ποσοστιαίες μονάδες είναι και εδώ σημείωτες με την Πολωνία και τη Σλοβακία να βρίσκονται κατά 20, να είναι σε 21 μονάδες ε, διαφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει στο 71% η Πολωνία, 78% η Σλοβακία. Και η Δημοκρατία της Τσεχίας, μην το ξεχάσω, είναι στις 90 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου στα επίπεδα της Ισπανίας. Να συνεχίσω σε κοινωνικούς δείκτες. Διότι όπως τα ξέρετε η πολιτική συνοχής αφορά και την οικονομική και την κοινωνική όμως συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το αποδεικνύει περίτρανα και επικεντρώνεται στο να φέρνει τον κόσμο στην αγορά εργασίας και να πιάνει δουλειά ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Πολωνία και η Σλοβακία όταν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν σε επίπεδα ρεκόρ ανεργίας. λόγω και των συνεπειών της μετάβασης από μια οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό σε μια οικονομία της αγοράς. Με ένα μεγάλο ποσοστό, 20% ανέργων ανθρώπων το 2014, η κατάσταση ήταν λιγότερο αρνητική στην Ουγγαρία εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά Ακόμα καλύτερη στην Τσεχία. 13 χρόνια μετά βλέπουμε ότι και η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν φτάσει στον ευρωπαϊκό μεσόωρο και με διαφορά ε, για την Πολωνία ειδικά ενώ η δημοκρατία της Τσεχίας είναι πρωταθλητής της χαμηλής ανεργίας. Είναι στο 2,4%. Βάσει των πιο πρόσφατων δεδομένων. Ο χαμηλότερο, το χαμηλότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία πέρασε από μια κατάσταση πολύ διαδεδομένης ανεργίας και με πολύ συγκεκριμένε ελλείψει δημοκρατικού δυναμικού σε συγκεκριμένου κλάδου πέρασε σήμερα σε ένα ιδιαίτερο άνοιγμα με εργάτες και εργαζομένους από την Ουκρανία. Εδώ και πάλι έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη από την προσχώρηση και μετά. Ένας ακόμη κοινωνικός δείκτης τώρα, το μερίδιο του πληθυσμού που απειλείται από την ένδυα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα στοιχεία μας αρχίζουν από το 2005 μόλις. Και πάλι η κατάσταση βελτιώνεται σε όλες τις χώρες. Πιο δραματικά είναι τα πράγματα στην Πολωνία. με 50% μείωση στο δίκτυ απειλής από τη φτώχεια. Τώρα είναι κάτω από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα που τα πηγαίνει λιγότερο καλά από αυτές τις τέσσερις είναι η Ουγγαρία που παραμένει πάνω από το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ η Δημοκρατία της Τσεχίας έχει τους χαμηλότερους αριθμούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που έχω ακούσει Τσέχους αξιωματούχους να διαφωνούν, θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ευρωπαϊκό ορισμό για την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό θεωρούν ότι παρουσιάζουμε πολύ πιο ρόδινη από την πραγματικότητα την εικόνα της Τσεχίας Παρ' όλα αυτά η κατάσταση κοινωνικά φαίνεται να είναι κάπως ομοιογενής ως προς τις δεξιότητες των εργαζομένων. Αν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε σημαντική πρόοδο. Εάν δούμε το μερίδιο του πληθυσμού μεταξύ 30 ε, και 34, 34 ε, ετών, δηλαδή στην τριτοβάθμια, στο τρίτο βαθμό, τριτοβάθμια εκπαίδευση, βλέπουμε το μερίδιο να έχει αυξηθεί εκρηκτικά με τριπλασια... τριπλασιασμό κάποιες φορές στη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία ας πούμε. Τρεις από τις τέσσερις χώρες του Βίζεγκραντ έχουν προλάβει τον ευρωπαϊκό μεσόρο κάτω από το 40% ε, τώρα, το 2017, και η Πολωνία έχει ξεπεράσει όλα τον ευρωπαϊκό μεσόρο με 45%. Βλέπουμε ωστόσο ότι όλα τα κράτη-μέλη πέραν της Ουγγαρίας έχουν επιτελέσει περισσότερη πρόοδο από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Αυτό είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, διότι μας δίνει και κάποιο, κάποια ιδέα για τη δυνατότητα ανάπτυξης στο μέλλον. Τα πρώτα στάδια όπου φτάνει κανείς στον ε, μέσο όρο των υπολείπων είναι τα πιο εύκολα. Με σταθερότερο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Αυτά προσελκύουν πολλές ε, ξένες άμεσες επενδύσεις και αυτά επιτρέπουν γοργή ανάπτυξη. Στην αρχή όλα τα κράτη-μέλη υποφελήθηκαν από αυτήν την αλλαγή. Τότε όμως φτάνει κανείς σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, οπότε εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες Εκεί αρχίζουν να χρειάζονται εργαζόμενοι με τις ψηλότερες δεξιότητες και εκεί αρχίζει να χρειάζεται περισσότερο καινοτόμος ανάπτυξη και μοντέλα πιο κοινοτόμου ανάπτυξης. Εδώ μπορούμε να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία που απαιτείται υπάρχει και διατίθεται σε αυτά τα κράτη-μέλη για να συνεχίσουν στην σωστή πορεία. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε συνοπτικά. Επόμενη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βλέπουμε συνοπτικά τι ισχύει ως φαινόμενο κατά κύριο λόγο επειδή ακριβώ αυτέ οι τέσσερι χώρε του Βίζεγκραντ έφτασαν στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με τον πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο που διδερματίζει η πρωτεύουσα ως αστικό κέντρο. Δηλαδή βλέπετε στη δημοκρατία της Τσεχίας οι περιφερειακές ανισότητες, ποιες ε, πώς διαμορφώνονται. Στην Πολωνία είναι πιο έντονο το φαινόμενο και στις άλλες δύο λιγότερο. Στις τέσσερις περιπτώσεις βλέπουμε την Πράγα, τη Βουδαπέστη, την Βαρσοβία και την Πρατισλάβα να έχουν φοβερή ανάπτυξη και να έχουν αναπτυχθεί γρηγορότερα από την υπόλοιπη χώρα από τον Εθνικό Μεσόρο. Στην Ουγγαρία βλέπετε ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν μειωθεί κάπως, δηλαδή η περιφέρεια της Βουδαπέστης έχει αναπτυχθεί κάπως βραδύτερα από την υπόλοιπη Ουγγαρία. Και αυτό δεν είναι κάτι το περίεργο. Είναι μάλλον αναμενόμενο. με τη γοργή ανάπτυξη πολλές φορές υπάρχει συγκέντρωση αυτής και θα ισχυριστώ εδώ πάλι ότι τα κονδύλια επέτρεψαν οι διαφορές αυτές, οι ανισότητες, να παραμένουν σε μια σχετική ισορροπία. Μπόρεσαν τελικά όλες οι περιφέρειες της χώρας να αναπτυχθούν ε, γοργότερα από ό,τι θα είχε γίνει χωρίς υποστήριξη. Επόμενη διαφάνεια. Πώς το πετύχαμε αυτό. Με εντυπωσιακού αριθμούς ως προς τη, τα κονδύλια της συνοχής. Και επίσης ένταση της βοήθειας ανακάτοικο ανακάτοικο-ανέτος σε αυτά τα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι το 2010, το 2007 έως 2013 η Δημοκρατία της Τσεχίας είχε τη μεγαλύτερη ένταση κατά κεφαλή από όλα τα κράτη-μέλη με την Ουγγαρία να ακολουθεί κατά πόδας. Η Σλοβακία είναι στην κορυφή μαζί με την Εστονία. Εδώ λοιπόν έχουμε τέσσερα κράτη-μέλη που και σε άποψη βάθος χρόνου έχουν λάβει τη μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εικοσαετία de facto και το λέω αυτό το de facto γιατί οι συνέπειες αυτής της περίοδου θα γίνονται στη τέσσερα το 2023 όπως έχουμε τον κανόνα N3 πολλές από τις επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν λάβει χώρα θα τις ε, ζήσουμε σε λίγο Βλέπετε ότι ως αναλογία του ΑΕΠ η σχέση, ο λόγος ήταν πολύ εντυπωσιακό. Η Ουγγαρία συστηματικά ελάμβανε περισσότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2017 το 2007 ως 2013 μία ποσοστία μονάδα παραπάνω από τις άλλες τρεις χώρες του Βίζεγκρατ και σε αυτή την τωρινή, την τρέχουσα περίοδο και πάλι λίγο παραπάνω από τους υπολείπους. Επόμενη διαφάνεια. Πώς θα πάνε αυτές, σήμερα αυτές, αυτές οι χώρες, στην τωρινή, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Έχουμε εδώ έναν δείκτη που ε, φωτίζει και τα υπόλοιπα στοιχεία. Η Ουγγαρία έχει αποδώσει τα περισσότερα κονδύλια της συνοχής σε συγκεκριμένα έργα και ως προς την εκτέλεση των προπολογισμών. Είναι στην κορυφή του καταλόγου της λίστας. Οι άλλες τρεις χώρες του Βίζεγκρατ είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο η Τσεχία και η Σλοβακία και πάνω από τον μέσο η Πολωνία. Η Πολωνία και σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού έχει σταθερές επιδόσεις στο ύψος των προηγούμενων και προοδεύει πολύ αρμονικά με καλή απορρόφηση των κοντιλίων αυτής της περίοδου. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ είναι κάπως λεπτομέρειες ε, αυτά που σας δείχνουμε. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε όλους αυτούς τους αριθμούς. Είναι μια κλασική παρουσίαση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την τρέχουσα περίοδο σε τομείς όπου ακόμη υποστηρίζουμε έργα όπως για υδροδότηση, για καθαρό νερό, για διαχείριση αποβλήτων, για τις υποδομές μεταφορών, για το ευρωζωνικό διαδίκτυο, για την υποστήριξη επιχειρήσεων. Αυτό όμω που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού και αυτό μας παραπέμπει σε ένα προηγούμενο σχόλιο μου για την ανάγκη βαθμιδών να αλλάξει η προσέγγιση για να συνεχίσουμε στον, στην πορεία της σύγκλησης αυτό λοιπόν που ισχύει είναι ότι για, και για τα τέσσερα κράτη-μέλη αυτά προοδευτικά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και καινοτομία. Με τα κονδύλια μας όλα αυτά τα κράτη-μέλη και τα τέσσερα θα βλέπουν το μερίδιο της έρευνας και καινοτομίας ως προς το ΑΕΠ τους να αυξάνεται σημαντικά ως το 2020. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη πορεία και έτσι την διαπραγματευτήκαμε και με αυτές τις τέσσερις χώρες. Και αυτή είναι και η δική μας συλλογιστική για την ερχόμενη περίοδο, δηλαδή βάσει των ευθειών στρατηγικών εξειδίκευσης θα δοθεί περισσότερη βαρύτητα στα προγράμματα έρευνας και κοινοτομίας, στα έργα υποδομών, στις δεξιότητες επίσης, διότι όπως θα είδατε η αγορά εργασίας των τεσσάρων αυτών κρατών μελών αρχίζει να στερεύει. Δεν υπάρχει περιθώριο. Πρέπει λοιπόν κανείς να επικεντρωθεί στην ε, αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Επόμενη διαφάνεια. Και τώρα να σας παρουσιάσω ε, κάποιες προσωμιώσεις βάσει των δικών μας μακροοικονομικών μοντέλων, αυτών που χρησιμοποιούμε στη Γενική Ρέτζη βάσει και του προτύπου της DG ECFIN. Εδώ προσπαθούμε να φωτογραφίσουμε, να απεικονίσουμε το καθαρό αντίκτυπο των επιπέδων του ΑΕΠ στις χώρες αυτές όπως προκύπτουν από τις δαπάνες της πολιτικής συνοχής. Εάν δούμε όλη αυτήν την περίοδο και το χρονικό σημείο που επιλέξαμε ήταν το 2017, δεν έχουμε ακόμα τις επιπτώσεις όλης της περίοδου πραγματισμού 2014-2020, Πιστεύουμε ότι θα πέσουν λίγο ρυθμοί το 2020, πάντως το 2017 και βάσει των προηγούμενων δαπανών συνοχής οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ως προς τα ΑΕΠ των τεσσάρων αυτών χωρών βρισκόμαστε σε, ποσοστίες, σε κάτι ποσοστίες μονάδες παραπάνω από αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε η πολιτική συνοχή, στην Πολωνία το ΕΠ θα ήταν 7% χαμηλότερο, της Ουγγαρίας 5% χαμηλότερο και της ε, Τσεχίας και Σλοβακίας 4% χαμηλότερα. Για να ολοκληρώσω. Ήθελα με κάθε σύνεση να ε, ισχυριστώ ότι η πολιτική συνοχής έχει εκπληρώσει τους βασικούς της σκοπούς να στηρίξει τις λιγότερα αναπτυγμένες περιφέρειες και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συγκλίνουν προς το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην περίπτωση αυτών των τεσσάρων κρατών μελών, χωρίς βεβαίως να ε, παραβλέπουμε ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία αυτών των τεσσάρων ή τέλο των τριών κρατών μελών ε, είχαν να κάνουν με την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Επίσης πρέπει να πω ότι για την πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτή τη θετική επίδραση στις οικονομίες των κρατών αυτών, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει στο μέλλον να επικεντρωθούμε περισσότερα στην καινοτομία και τις δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Δευτά. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είναι από τις καλύτερες μέρες μας. Και το χειρότερο θα ήταν να μας δώσετε κάποια στοιχεία μόνο και να μας πείτε ότι ε, είναι 260 τα δις και τα λοιπά και τα λοιπά και πώς θα έχουμε ε, διασπεί. Έχουμε λοιπόν αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται μια παράληψη να πω ότι για πρώτη φορά έχουμε εδώ τον κύριο Μέρφε ως μέλος της ε, συνάντησης μας στο Ευρωπαϊκό Ελληνικτικό Συνέδριο. Κυρία Λαμπάγιοβα, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, πάντοτε είναι καλή στιγμή, το είπατε και εσείς στην αρχή, να κάνουμε ένα βήμα πίσω ε, και να δούμε τους σημαντικούς αυτούς ε, στόχους ε, και τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Αυτό που έμαθα εγώ είναι πρώτον ότι δεν είναι τίποτα ασπρομαύρο, ακόμη και για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Οι καλύτεροι μπορεί να γίνουν χειρότεροι και το αντίθετο. Και επίσης ε, ότι βλέπουμε η Κομισιό να μπορεί να μας δίνει αξιόπιστα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό πάντοτε ζητούσαμε και στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας ε, απαλλαγής. Ξέρετε ότι ψηφίσαμε χθε μάλιστα για την απαλλαγή της Επιτροπής. Στην Επιτροπή μας δώσετε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι κάτι το οποίο εμεί ζητούσαμε. Θέλαμε να δούμε ποιο είναι ο πραγματικό αντίκτυπο πολιτική συνέχεια. Σα ευχαριστούμε λοιπόν. Είναι πολύ καλό επίση να αναφέρονται κάποιε φορέ οι καλέ βέλτιστες πρακτικέ, συγκεκριμένα έργα και προγράμματα θετικά. επιτυχημένε ιστορίε για την Τσεχία από την Υπουργείο Ανάπτυξη, ε, χάρη, υπάρχει ένα χάρτη ε, των προγραμμάτων και βλέπει κανεί τον αντίκτυπο, τα ε, έργα αυτά πώ επηρεάζουν και ποια είναι η προσθέμενη αξία του. Έρχομαι στην προσθέμενη αξία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε ποια είναι τα πραγματικά ωφέλη της πολιτικής συνοχής. Πολλά από αυτά τα αναφέρατε και μας δώσετε και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Έχω όμως ένα φιλοσοφικό ερώτημα για να έχουμε μια συνέχεια σε αυτά. Δεν ωφελήθηκαν μόνο οι τέσσερι σημαντικοί δικαιούχοι, αλλά η Ένωση συνολικά ωφελήθηκε από τι επενδύσει και από την πολιτική συνοχή. Μιλάγαμε για την προσθέμενη αξία ε, εντόνως τελευταία, την ευρωπαϊκή προσθέμενη και τη βλέπουμε. Σε διάφορα και αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα διάφορα. Ένα είναι η πολιτική συνοχή, που πιστεύω ότι είναι η πραγματική προσθέμενη αξία ουσιαστικά. Με μεμονωμένα τέτοια προγράμματα μπορεί να μην είχαμε την προσθέμενη αλλά συνολικά όλα τα προγράμματα έχουν πολύ μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Άρα νομίζω ότι το πακέτο αυτών των project θα έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειώνοντα, για παράδειγμα, τι περιφερειακέ ανισότητε, αυξάνοντα την απασχόληση, βελτιώνοντα το φοιτικό επίπεδο, την προστασία του περιβάλλοντο και άλλα. Και... Συμφωνώ, όπω είπατε και εσεί, ότι χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική συνοχή και στο προσεχέ πι. Το βλέπουμε όμω αυτό από τα απορίσματα και τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία. Αυτή είναι η αξία για την οποία μιλάμε. Ευχαριστώ πάντως για την παρουσίαση γιατί κάποια στοιχεία για μένα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια δεν τα ήξερα. Ελπίζω να είστε παράδειγμα καλό και για άλλους γενικούς διευθυντές. Να έρχονται με αντίστοιχα δεδομένα στην Επιτροπή Λεκτού Προϋπολογισμού. Κύριος Στεχόφσκι. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για την εντυπωσιακή παρουσίασή σας Πράγματι με εντυπωσίασαν οι αριθμοί και τα σχόλιά σας. Και αν στην τσεχική δημοκρατία μπορείτε να έρθετε και να μας δώσετε όλους τους αριθμούς θα ήταν πολύ καλό. Όντως έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τα παρατηρήσεις σας. Το ερώτημά μου αφορά την Επιτροπή μας και τους λέγχους που γίνονται εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι θέλουμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να χειριζόμαστε όλα αυτά τα θέματα με τον καλύτερα δυνατό τρόπο. Ε, μιλήσατε για το ΑΕΠ κάποιων χωρών. Έχω εδώ κάποια στοιχεία στα εγχειρίδια αυτά για να δείτε ποιες είναι οι δικές μας επιτεύξεις και να τις ε, συγκρίνετε με άλλες χώρες. Πολλές εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες προέρχονται από χώρες της Δυτικής, πρώην Δυτικής και Νότιας Ευρώπης. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Πολλά <coughs> project τα παίρνουν κάποιες αδιαφανείς επιχειρήσεις. Πολλοί δεν γνωρίζουμε και κανείς ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις ποια είναι η δομή τους, ποιος κρύβεται από πίσω. Από πού προέρχονται, από τη Ρωσία, από κάποια άλλη χώρα. Και θέθηκε το θέμα για όλες τις χώρες μας. Θέλω λοιπόν να σας ερωτήσω, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερο. Υπάρχουν και διάφορες έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για κάποια ειδικά προγράμματα. διότι κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν χρήματα από τα Ταμεία Συνοχής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάτε εσείς για τους ελέγχους που κάνετε. Είπατε ότι κάνετε πολλούς ελέγχους. Αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα κατά την γενική σας διεύθυνση. Εάν συγκρίνω τους ελέγχους που κάνετε με τα πορίσματα στα οποία καταλήγει ο ΟΛΑΦ, Πολλέ φορέ λέτε μετά από έναν έλεγχο δεν συνέβη τίποτα, ενώ είναι διαφορετική η ερμηνεία που δίδεται από την ΟΛΑΦ. Προβλέπετε κάποιες αλλαγές στο μέλλον, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και των ελέγχων που κάνετε. Ευχαριστώ. Εμείς ήσασταν εδώ σε μια συζήτηση που Μιλήσαμε για κάποιες παραλήψεις και κατάχρηση ε, στην, της, των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για τη Σλοβακία, την ε, Ουγγαρία, την ε, Πολωνία. Μας απασχολεί αυτό το θέμα. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά. κυρία Ζόντροβα, επόμενη. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι δεν με εκπλήσει ο θετικό αντίκτυπο για τον οποίο έκανε λόγο ο Γενικό Διευθυντή. Είμαι πεπισμένη ότι τα κονδύλια τη συνοχή επηρεάζουν θετικά την Τσεχία, για παράδειγμα, συγκεκριμένα, και το γνωρίζω γιατί έρχομαι από μια περιφέρεια που έχει αξιοποιήσει πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια από την Ανατολική Τσεχία συγκεκριμένα. Χωρίς αυτά τα κονδύλια συνοχής θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η ε, κατάσταση και δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά ε, το ποσοστό απορρόφησης, αυτό νομίζω ότι οφείλεται στις αλλαγές, στα Υπουργεία και σε κάποια στάθεια στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Είδαμε επίσης και στα γραφήματα ότι υπάρχουν πόροι που διατίθενται για την αύξηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Είπατε ότι πλέον το βάρος πέφτει στην έρευνα και την ανάπτυξη. Συμφωνώ, όμως θέλω να παρατηρήσω το εξής. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις ε, ανισότητες μεταξύ περιφερειών ή μεταξύ πρωτεύουσα και ε, αγροτικών περιοχών, γιατί οι περισσότερες δραστηριότητε, έρευνα και ανάπτυξης γίνονται στην, ε, στις μεγάλες ε, πόλεις, Πράγα, τον Πρνό και εκεί είναι η κινητήρη, η μοχλή της ανάπτυξης. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν πιο βαθιές οι ανισότητες μεταξύ των μεγάλου πόλεων και άλλων περιοχών, αν επενδύσουμε μόνο σε αυτές τις υποδομές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις υποδομές γενικότερα στις περιφέρειες. Ευχαριστώ κύριο Λιμπεράτσικη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν μπόρεσα να ακούσω την παρουσίαση. Διότι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχα άλλε υποχρεώσει ανηλυμένε, αλλά εν πάση περιπτώσει σα ευχαριστώ για την παρουσίαση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό από την οπτική γωνία της πολιτικής συνοχής είναι να δούμε πόσο εκτελούνται τα διάφορα προγράμματα. Βλέπουμε πολλές φορές ότι διάφορα ε, προγράμματα που ασχολούν έργα υποδομής αρχίζουν, γίνεται η πρώτη φάση τους και δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και βεβαίως θα είναι καλύτερη η συνοχή εάν φέρει πίν ένας αυτοκινητόδρομος γίνεται εξ ολοκλήρου και με ενιαίο τρόπο από τη μια μεριά των συνόρων μέχρι την άλλη. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα κονδύλια εξαρτώνται από πολιτικές ε, ε θεωρήσεις, ε, κατακαιρματίζονται κυρίως για τα οδικά έργα και δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι υπολείπονται στην Πολωνία Φερι, θα αναφέρω τη έργα υποδομής των σιδηροδρόμων, τα οποία πραγματικά υπολείπονται άλλων υποδομών. Και δεν υπάρχει αρκετή πίεση ώστε τέτοιου είδους προγράμματα να προχωρήσουν. Έχει λοιπόν μία, έχει εκφράσει μία κάποια έχει επιδείξει ένα κάποιο ενδιασμό η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια θέματα τέτοια. Και ίσως πολλές φορές είναι και θέμα εμπορίας. Κάνετε τούτο για να κάνουμε το άλλο. Ε, πάρτε από εκεί τον εξοπλισμό για να προχωρήσει κάτι άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους προγραμμάτων υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ πιο αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρόκειται για τέτοιου είδους προγράμματα. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να μιλούμε για πραγματικά προστιθέμενη αξία σε αυτά τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υπάρχουν ε, περιοχές στις οποίες ε, έχουν περισσότερη επιρροή από άλλες ή έχουν περισσότερους πολιτικούς κτλ. Εδώ παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή μας τα παραδείγματα για τους πολωνικούς σιδηροδρόμους ως κάτι το αρνητικό. Θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενεργεί σε τέτοιου είδου θέματα. Μήπω θα έπρεπε η Επιτροπή μα να κάνει κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάμπον. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενημερωτική παρουσίαση που αφορά τις επιδόσεις στα πλαίσια τη πολιτικής συνοχής των χωρών Βίσιγκραντ. Υπάρχει μια κάπως αρνητική εικόνα για τη χώρα μου την Ουγγαρία που φαίνεται ότι είναι εξαίρεση σε σχέση με άλλες χώρες. Το γνωρίζουμε αυτό από καιρό και προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η εξήγηση. Υπάρχει πρόοδο στην Ουγγαρία, κύριε Λεμέτρα. Ίσως κάτι δεν ε, υπάρχει σαφώς στην ομιλία σας. Υπάρχει σαφής εικόνα για να, δείξουμε, για να δείξετε γιατί είναι διαφορετική από τι άλλε χώρες η Ουγγαρία. Για ποιο λόγο. Τι δεν πάει καλά στην Ουγγαρία με όλα αυτά τα κοινοτικά κονδύλια στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής. Η διαφθορά, έχουμε υψηλότερο ποσοστό διαφθοράς, γι' αυτό οι επιδόσεις μας δεν είναι καλές στην Ουγγαρία. Μήπως ε, ε, Εξαιτία πολιτικών ε, ε, θεωρήσεων, όπως είπε και ο συνάδελφος, κατασπαταλώνται κάποια κονδύλια και δεν καταλήγουν πουθενά τα προγράμματα. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις για να δούμε γιατί αποτυγχάνει σε κάποια κράτη-μέλη πολιτική συνοχή και τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις χώρες αυτές και να τις υποχρεώσει να χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια καλύτερα. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε την ε, διαφθορά. Μπορεί να βοηθήσει η Επιτροπή να προκάνει κάποιες προτάσεις ή θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει οι κανόνες ε, που πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο αυστηρή ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Διαφορετικά και στις επόμενες χρονιές, όπως κάναμε μέχρι τώρα, πολλές ε, φορές τα πλαίσια των ε, νομοθετικών κύκλων που ορίζουμε, θα συνεχίσουμε να πετάμε κάποια χρήματα και να τα κατασπαταλούμε. Θα θέλαμε λοιπόν για όλες αυτές τις διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών να μας δώσετε σαφέστερες εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ πιστεύω ότι η υποστήριξη μέσω των κορδιλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, επέφεραν πολύ σημαντικές αλλαγές. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι για χρόνια και δεκαετίες Μιλάμε για κράτη που ε, ήταν σε περίοδο μετασχηματισμού, δηλαδή από το 1990-1991 είχαν ε, αλλάξει εντελώ το μοντέλο, το σοσιαλιστικό κολυβιστικό μοντέλο, όπου υπήρχε ένα και μόνο κόμμα το οποίο ε, κανόνιζε και η αρχή του Μάρξ ο άνθρωπος είναι το κεφάλαιο καθόριζε την πολιτική με την κατάργηση ε, του σοσιαλισμού και την εισαγωγή στοιχείων οικονομίας της αγοράς. Υπήρξαν ε, πολλές εταιρείες από τη Δύση που καταστάθηκαν ε, στις χώρες αυτές για να έχουν κέρδη και πράγματι είχαν πολλά κέρδη αρχικά. αλλά ε, όλα αυτά ωφέλησαν ε, και τις παλιές κομμουνιστικές ελίτ που ήξεραν πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ε, την κατάσταση που είχε. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις την επίδραση αυτής της ελίτ τη βλέπουμε ακόμη και επηρεάζει και την ανάπτυξη. Υπάρχουν παράπονα τα οποία έχουν εκφραστεί σήμερα σε σχέση με κάποια ζητήματα όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις και που είναι ανησυχητικά. Βέβαια ελπίζουμε ότι υπάρχει πλέον και αυτή η κοινωνία των πολιτών που αναπτύσσεται και που παρακολουθεί ε, αυτούς ε, που ε, πλουτίζουν και κερδοσκοπούν. Το πώς βέβαια ε, αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο το είδαμε στην Σλοβακία, το είδαμε και στη Μάλτα που μια δημοσιογράφος δολοφονήθηκε γιατί είχε έρθει στα ίχνη κάποιων που παρανομούσαν και έκαναν καταχρήσεις. Είδαμε τα στοιχεία από την Πολωνία και από τις άλλες χώρες και αυτά τα θετικά στοιχεία ακριβώς ε, είναι τόσο θετικά γιατί είναι μέλη της Ένωσης οι χώρες αυτές. Υπάρχει μια μετακίνηση εργατικού δυναμικού. Έχουμε την ε, μετακίνηση πάρα πολλών Πολωνών ε, Παραδείγματο χάρη στη, το ένα στα δύο αυτοκίνητα έχουν πολωνικές πινακίδες στη χώρα μου και στο Βερολίνο έχουμε πάρα πολλούς ε, υπηκός Πολωνίας ε, που έχουν έρθει και εγκατασταθεί. Υπάρχει λοιπόν η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Το είπε και ο κύριος Λεμέτρο. Υπάρχει βέβαια έλλειμμα στις χώρες αυτές από τις οποίες φεύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι για να έρθουν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Υπάρχει φυγή ε, πολλών εργαζομένων από την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ιδίως για τις ε, χώρες αυτές. Για πείτε μας, αν και εσείς είστε ικανοποιημένος 62 ε, δις δεν είναι και μικρό ποσό. Κύριε Λεμέτρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις. Δεν πρέπει να είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον αντίκτυπο που έχουν οι δημόσιες δαπάνες και ιδίως οι δαπάνες για επενδύσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία των συναδέλφων στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΓΙΟ. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε ακόμα ανακαλύψει ε, τη μαγική φόρμουλα για την ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι το έχει καταφέρει κανείς στον κόσμο αυτό. Και πάντοτε μαθαίνουμε. Γι' αυτό και Χαίρομαι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να σκεφτούμε λίγο όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μία πολύ ανοιχτόμυαλη προσέγγιση. Θέλουμε να βρούμε καλές πρακτικές και καλά συστατικά για το μέλλον. Αυτό το βλέπετε και στα πολλά πιλωτικά προγράμματα που έχουμε δρομολογήσει μέσα στα τελευταία χρόνια. Ιδίως για τις περιοχές που απέχουν περισσότερο από το μέσο όρο, τον ευρωπαϊκό. Και που ίσως μείνουν πίσω, όπως είπατε. αν μόνο οι πρωτεύουσε αναπτύσσονται. Έχουμε την, προπο, την τροπολογία για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε υστέρηση, lagging regions initiative. Μαθαίνουμε από τα πειράματα αυτά. Νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία που μας εμπνέει και έτσι προχωρούμε χωρίς σε καμία περίπτωση να υποστηρίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αντίθετα, είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας πείσω ότι δεν είμαστε απαθείς μπροστά σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη, γιατί φάνηκε από τις ερωτήσεις σας ότι δεν έχετε, δεν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι προσέχουμε την κατάσταση. Όχι, προσέχουμε πάρα πολύ την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Για να μην μακρηγορήσω, περνάω στις ε, ερωτήσεις. Κυρία Αντλαμπάγιοβα. Ναι. Πράγματι, τα ωφέλη στα μεμονωμένα κράτη-μέλη δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Είναι προφανές ότι οι πολύ θετικέ εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα που σας περιουσίασα ωφελούν και άλλα κράτη-μέλη μέσω της ενές αγοράς. Και θα έλεγα με δύο τρόπους. Μέσω των συμβάσεων που ανατίθενται Πολλές αδετικές εταιρείε ε, έχουν ε, πάρει συμβάσεις ε, για έργα υποδομών. Δεύτερον, αυτή η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό και την ανάπτυξη του εμπορίου. όπως απεικονίζεται στο μερίδιο των εξαγωγών που έχει αυξηθεί για τις χώρες αυτές αυξημένο εμπόριο, το οποίο ωφελεί βέβαια και πάλι όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. right Υπάρχει και ένα ακόμη σημείο στα διάταξη. Το επόμενο συγκεκριμένο που αφορά μια συγκεκριμένη τσεχική εταιρεία. Ο κύριος Τσεχόφσκι όμως ήδη έθεσε σχετικά ένα ερώτημα. δηλαδή την αδιαφάνεια. Αδιαφανείς εταιρείε που ωφελούνται από κάποια έργα. Και τι θα κάναμε. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια γενική απάντηση. Για χρόνια είχαμε στην Τσεχική Δημοκρατία το φαινόμενο να επιτρέπονται οι υποβολές προσφορών από ανώνυμους υποψηφίους αναδόχους και μπορούσε να είναι άγνωστο ο διοκτήτης της εταιρείας. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο ζήτησαν ψυχή δημοκρατία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συστάσεις ε, εδώ και χρόνια και τώρα με τέταρτη οδηγία για την νομοποίηση εσόδων παρών δραστηριότητες που έχει μεταφέρει στο Εθνικό Δίκαιο από την Τσεχία Έχουμε λοιπόν τώρα με αυτή την οδηγία θετικές εξελίξεις. Οι ανώνυμοι μέτοχοι δεν είναι κάτι το οποίο πλέον επιτρέπεται στην Τσεχική Δημοκρατία. Άρα μπορούμε να ησυχάσουμε. Όχι εντελώς όμως, όχι εντελώς, διότι οι διαχειριστικές αρχές όταν υπάρχουν ειδικά προγράμματα που αφορούν, αποφθύνονται σε ΜΜΕ, διαχρηστικές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν ότι πρόκειται πραγματικά περί ΜΜΕ. Όταν κάναμε ένα συστημικό έλεγχο στη Τσεχία πριν από ένα χρόνο, δεν μας ικανοποίησε πλήρως ο τρόπος με τον οποίο ενερευνούσαν τις πληροφορίες που έδιναν οι εταιρείε οι αρχές δεν σκάλιζαν σε βάθος. Ζητήσαμε λοιπόν από τις διαχειριστικές αρχές να προβαίνουν σε συστηματικούς ενδελεγείς ελέγχους, κάτι το οποίο κάνουν τώρα. Ένα άλλο γενικότερο ερώτημα ήταν ποιοι είναι σημεία επιπτώσει των ελέγχων. Αν δείτε την τελευταία περίοδο, με τους ελέγχους μας, είχαμε δύο δις διορθώσεις. Και συνολικά, το σύστημα δείξε περισσότερες διορθώσεις από το εθνικά συστήματα. Ήδη λοιπόν σας έχουμε στείλει τέτοια στοιχεία και αν θέλετε μπορούμε να σας ξαναστείλουμε. Σε αυτό το μέτωπο και εδώ μιλάμε για τα ασφάλματα, έχουμε νομίζω καταδείξει και είμαστε και στη διαδικασία που με τη διαδικασία κλεισίματος που συνεχίζεται για το 2013 συνεχίζουμε να καταδεικνύουμε ότι το ποσοστό πολυματικού σφάλματος θα είναι κάτω από 2%. Απάτη. Γιατί νομίζω ότι γι' αυτό μιλούσατε όταν αναφερθήκατε στις εκθέσεις της Όλαφ. Ναι, πράγματι. δεν καταλήγουν πάντα στα ίδια συμπεράσματα. Με την Όλαφ, η εκθέση της Όλαφ υποβάλλονται συστηματικά σε εθνικές αρχές. οι εθνικές αρχές μπορούν στη συνέχεια να απαντήσουν, να αντιδράσουν παρέχοντας ενδεχομένω πρόσθετες πληροφορίες και το καθεξής. Και αυτό πολύ συχνά οδηγεί σε διόρθωση, αλλά ίσως όχι στο 100%. της προτινόμενης από την Όλαφ διόρθωσης, τουλάχιστον κατά το παρελθόν. Πάντως, Παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά τις εκθέσεις της Όλαφ και το πώς οι συστάσεις της εφαρμόζονται. Δηλαδή αν έχουν διορθωθεί τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν και ούτω καθεξής. Δεν είναι όμως μόνο η απάτη, για την απάτη σίγουρα μιλάμε για 100% και όχι πιο κάτω, με διόρθωση κυρία Είπατε κι εσείς ότι ίσως δεν έχει αναπτυχθεί τόσο θετικά η τσεχική δημοκρατία όσο θα έπρεπε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Το διαπιστώνουμε αυτό, αλλά Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Θα πρέπει ίσως να επικεντρωθούμε ίσως άλλα θέματα και ίσως τα θέματα της κοινοτομίας να οδηγήσουν ίσως σε μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να το προστέξουμε το θέμα αυτό. Τα έργα υποδομής δεν είναι η μοναδική λύση για να ανακτήσει κάποιος την καθυστέρηση σε κάποιους τομείς. Η καινοτομία πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την ε, ευφυή προσέγγιση που έχουμε σε όλα αυτά τα θέματα και σε συνεργασία με τις αρχές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο γιατί προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε ποιες είναι, ποια είναι τα δυνατά του σημεία για να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο για να προχωρήσουμε. Γενικότερα θα ήθελα να πω το εξής. Βλέποντας όλες αυτές τις πολύ θετικές εξελίξεις προς ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τάσεις που διαγράφονται όσον αφορά τα κονδύλια αυτά που διατίθενται στις τέσσερις χώρες αυτές τα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, αλλά και εκείνες θα πρέπει να δουν ε, με πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα αυτή την ε, υποστήριξη την οικονομική, η οποία όμως ε, αναμφίβολα σιγά σιγά θα αρχίσει να μειώνεται. Κύριε Λιμπεράτσκι, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Πρωτοπολώς, όσον αφορά τα ατελή, τα ημιτελή προγράμματα. Εάν δεν ολοκληρώνονται και αν δεν είναι λειτουργικά τα project αυτά, θα πρέπει να υποστραφούν τα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή σας, όντως, πάρα πολύ εμπεριστατωμένα έχει εξετάσει το άλλο θέμα, διότι υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις και μετά από την περίοδο χάριτος που δίδουμε, πάντα εξετάζουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και μετά από το Μάρτιο του 2009 θα δούμε τι έχει ολοκληρωθεί, τι λειτουργεί ή όχι. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς. Τα project όχι μόνο πρέπει να ολοκληρωθούν, αλλά και να τεθούν σε εφαρμογή, σε ισχύ. Για να συνεχίζει να παρέχεται υποστήριξη. Αναφέρατε το παράδειγμα των αυτοκινητοδρόμων που δεν ολοκληρώνονται από τα βόρειο τα νότια σύνορα της χώρας, από τα ανατολικά στα δυτικά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Προφανώς οι αυτοκινητόδρομοι παντού στην Ευρώπη ολοκληρώνονται σταδιακά και κατακαιρματισμένα. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα για 20-30 χιλιόμετρα και μετά συνεχίζονται. Δεν είναι διαφορετική η πολιτική που ακολουθείτε στη χώρα σας και βεβαίως γίνονται κάποιες επιλογές από τις κυβερνήσεις που αποφασίζουν ποιο κομμάτι θα ολοκληρωθεί πρώτα για λόγους χρησιμότητας, για λόγους ευκολίας, εν πάση περιπτώσει. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι μιλάτε για την A6 στην Βόρεια Πολωνία. Επιμείνουμε στο ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί ώστε το η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία αυτού του έργου να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά τις σιδηροδρόμους και τα έργα υποδομής. Διαφωνώ με την δική σας την εκτίμηση. Εγώ πήγα στην Πολωνία για την ε, δημιουργεί και θέσει λειτουργία μιας κοινή task force μεταξύ της κυβέρνησης, των πολωνικών ε, σιδηροδρόμων σχετικού οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την συνδρομή και της Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να ασκηθεί όσο περισσότερη πολιτική πίεση μπορεί να ασκηθεί, ώστε να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να έχει καλές επιδόσεις, γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Ποιος ήταν ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι τα δισεκατομμύρια που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την περίοδο, ναι, να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι αληθές ότι στην προηγούμενη περίοδο, σε σχέση με τα αρχικά στάδια, υπήρχε μια κάποια ε, αλλαγή σε σχέση με τη βελτίωση των ε, δικτύων. Και αντικαταστάθηκε ένα μέρος του τροχαίου υλικού, ίσως γιατί δεν υπήρχε οριμότητα στα σχετικά ε, προγράμματα που αφορούσαν το δίκτυο. Και βεβαίω ήταν πολύ πιο ελκυστική η αντικατάσταση του τροχαίου υλικού, πράγμα το οποίο φαίνεται από την αύξηση των ατόμων που χρησιμοποιούν του σιδηροδρόμους. Αύξηση, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, του 40% τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. Βεβαίω δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση και δεν θα μείνουμε εδώ. Αλλά θα προσπαθήσουμε και να βελτιώσουμε και γενικότερα το δίκτυο, αλλά και με την βοήθεια της Task Force αυτής και είναι μαζί μας η υπεύθυνο για το θέμα αυτό που το παρακολουθεί εξάλλου. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις και μπορώ να σας πω ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με την πολωνική κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί ο στόχος μας και να επιτευχθεί πρόοδος. Όσον αφορά τώρα την κατανομή κονδυλίων για project με των διαφόρων προγραμμάτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Πολωνίας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού τα κονδύλια κατανέμονται ανά περιοχή σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% από το περισσότερο λοιπόν το 50% των σχεδίων αφορά περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος προγράμματα και δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Βεβαίως, εστιάζουμε την προσοχή μας περισσότερο στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά αυτό έχει μια κάποια αιτιολόγηση. Αν δείτε ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης στην περιοχή σας, θα δείτε ότι αυτές είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Σήμερα στην Πολωνία υπάρχουν περιοχές, περιφέρειες, οι οποίες περίπου βρίσκονται στο 50% του μέσου κοινοτικού όρου. Τελικά, κύριε Μπερναντέκ. Γιατί η Ουγγαρία δεν τα πήγε τόσο καλά όσο οι άλλες χώρες μέλη. Όντως, περί αυτού πρόκειται. Αλλά έχουμε υποεξέταση μία περίοδο η οποία έχει ιδιαιτερότητες, δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνει την πιο σοβαρή οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη εδώ και 8 χρόνια. Και βεβαίως οι επιπτώσεις για την Ουγγαρία ήταν πολύ πιο σοβαρές από τις Άλλε χώρε. Αν δεν κάνω λάθο υπάρχουν πιστώσει με τα οποία εποφελούνται ε, τα προγράμματα τη χώρα σα τα οικονομικά και από εμά και από το νομισμα... Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ε, οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας υπέφερε και υποφέρει από αυτή την κατάσταση και το δείχνουν και οι γραφικές παραστάσεις που σας παρουσίασα. Επίσης, μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα πάει κάπως καλύτερα η Πολωνία σε σχέση με τους άλλους, τις τρεις χώρες και αρχίζει και, αρχίζει και παρουσιάζει καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Στα πλαίσια τώρα των συστάσεων για τις χώρες αυτές. Η Ουγγαρία είναι διαφορετική. διότι είχε μεγαλύτερη αναλογία ε, δημοσίων δαπανών από ό,τι οι άλλες χώρες, σε ποσοστά παρεμφερεί με τις περισσότερες ανεπτυσμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε ποσοστό 50% και δεν ήταν ε, και πολύ επιτυχής δεδομένης αυτής της ασταθούς μακροοικονομικής κατάστασης. Όσον αφορά την προσέλκυση κονδυλίων σε σχέση με τις άλλες τρεις χώρες. Επικεντρωθήκαμε όμως αυτή την περίοδο και προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα διάφορα κονδύλια σε τομείς καινοτόμους και η Ουγγαρία ξέρουμε ότι για έργα έρευνας και ανάπτυξης από το 1,3 θα φτάσει το 2020 στο 1,8, πράγμα που είναι αξιοσημείωτο ως ε, διαφορά, ως αύξηση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα κονδύλια μας θα έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην μακροοικονομική προσωμείωση την οποία σας έδειξα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά στα πορίσματα στα οποία καταλήξαμε στην ε, Ουγγαρία. Όπως είπα, ίσως υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα γενικότερα της Ουγγαρίας. Και οι επιπτώσεις βεβαίως αυτές ανέρχονται στο 5 1,3% του ΑΕΠ το 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της περίοδου που εξέτασε. Ευχαριστώ. Κύριος Μέρφη, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και για την ευκαιρία να ακούσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική συνοχή που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μένα. Διότι είμαι υπεύθυνο για το σχετικό κεφάλαιο στην ατήσια έκθεση. Όπως είπε ο κύριος Λεμέτρα στην παρουσίασή του, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της χρηματοδότηση από τα Ταμεία Συνοχή και της ανάπτυξη στα κάτι Είναι σημαντικό ο πολιτικό κλάδο αυτό. Γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάνει πολλή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Με πολλού ελέγχου και το κεφάλαιο είναι η κατάληξη που ανέφερα με ειδικέ εκθέσεις που επίσης υποβάλλονται στην Επιτροπή σας και πολύ σύντομα λίγα λόγια για τη δράση του ελεγκτικού συνεδρίου προς τους ελέγχους για την πολιτική συνοχή. Η νομιμότητα και η νομοτυπία είναι θέματα που μας απασχολούν κάθε χρόνο για να εκτιμήσουμε τις επιδόσεις της πολιτικής συνοχής συνολικά ανάλογα με τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Για το επίπεδο σφάλματος ε, που ήταν υψηλότερο στο παρελθόν, είδαμε μια τάση μείωση του ποσοστού αυτού από το 2007 σε 11% σε 4,8% το 2016. Είναι λοιπόν μια προσδεκτή εξέλιξη. Παρόλα αυτά είναι ακόμη πάλι από το επίπεδο του ενότερο επιτρεπτό του 2% και πρέπει να το διορθώσουμε κι άλλο. Επίσης, ξέρουμε ότι τα προγράμματα και οι επιδόσεις τους ως προς την ε, συνοχή και τις δράσεις που αφορούν τη συνοχή, το 2018 είχαμε μεγάλες, ε, μεγάλους ελέγχους για την απλούστευση της πολιτικής συνοχής, ελέγχους προτεραιότητας και αυτό θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει στη συζήτησή σας. Δύο άλλα σημεία που θέλω να αναφέρω είναι ότι το 2015 είχαμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό μάλλον έλεγχο για τους διαγωνισμούς και μετά για τη Βουλγαρία, Λετωνία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Γαλλία κλπ. Επτά κράτη-μέλη συνολικά κάναμε έλεγχο για τη διαφθορά στους διαγωνισμούς και θα το ξανακάνουμε και το 2019. Προ στιγμή καταρτίζουμε το πρόγραμμα εργασιών μα για το 2019, όπου θα σκεφτούμε και άλλε προτάσει από διαφορετικού εταίρου, μεταξύ των οποίων η ε, διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και η διάσκεψη των Προέδρων και πάλι μπορεί να μελετήσουμε και άλλες πτυχές των δημόσιων προμηθειών σε σχέση με το 2015. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που ήθελα να υποβάλω και να σας αναφέρω σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο της διάταξης. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, πρέπει να παραμείνετε για το επόμενο ε, σημείο που είναι η παρακολούθηση του έργου Storks Nest. Ζητήθηκε να μην γίνει και κλεισμένο των θυρών ε, το, η συζήτηση του θέματος γιατί είναι γνωστό τη Πάσιν. Οπότε έχετε το λόγο να μας δώσετε τα σχόλιά σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα παρουσιάσω χρονολογικός. Το Μάρτιο του 2017, όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη έπρεπε να μας υποβάλουν ε, τα πακέτα κλεισίματος για τα προγράμματα της περίοδου 2007-2013. Η τσεχική δημοκρατία το έπραξε δεν των αρχών της ε, και για το πρόγραμμα ναι, που αφορούσε την κεντρική βοημία και στο οποίο περιλαμβανόταν μια υποστήριξη 2 εκατομμύρων ευρώ περίπου σε μια εταιρεία ονόματι Stork Nest, φωλιά του πελαργού. Οι αρχές εν συνεχεία μας είπαν ότι το είδος αυτό, τη δαπάνη συγκεκριμένη στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος θα ερευνά το διότι υπήρχαν ε, και έρευνες από την Όλαφ και την αντίστοιχη αρχή στη χώρα. Τον πέρσινο Δεκέμβρη η Όλαφ ολοκλήρωσε την έκθεσή της, την οποία και λάβαμε. Στην έκθεση αυτή, μάλλον την έκθεση αυτή τη διαβάσαμε στις τσεχικές αρχές και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν μία ανεξάρτητη ΜΜΕ η φωλιά του πελαργού, αλλά εντασσόταν στον όμιλο Άγκροφερτ. Άρα δεν ήταν επιλέξιμη για στήριξη σε ΜΜΕ. Με βάση λοιπόν τα συμπεράσματα της Όλαφ, προτείναμε στις εκεί αρχές να αποσύρουν τη δαπάνη από το πρόγραμμα για την κεντρική βοημία. Όπερ και δέχτησαν, με το Φεβρουάριο. Οπότε μπορέσαμε μετά να προχωρήσουμε στο κλείσιμο του προγράμματος. Με την αφαίρεση αυτού του προγράμματος. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Δεν δόθηκε δηλαδή υποστήριξη από τον Ευρωπαϊκό Περιπολογισμό σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σημαντικό. Αυτό που μας είπατε, σημαντική διευκρίνηση, ο οποίος Στεχόφσκι. Ευχαριστούμε Γενική Διευθυντά για αυτή την ε, εξήγηση. Διάβασα την έκθεση της Όλαφ, η οποία διέρευσε μου είπαν επανειλημμένος ότι θα γίνει επίσκεψη στις ε, Βρυξέλλες για να δοθούν εξηγήσει. Πάντως καμία επίσημη δράση δεν αναλήφθη κατά του Πρωθυπουργού Μπάμπης. Το ερώτημα είναι πώς συνέβη αυτό και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση στο μέλλον. Εάν διαβάσετε την έκθεση της Όλαβ στο προήμιο, βρίσκονται πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δηλαδή ότι η εταιρεία ευθύ εξ αρχής δεν ε, ήταν διαφανής, κανείς δεν γνώριζε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης Και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να ιδρύει κανεί εταιρεία και να διεκδικεί διαγωνισμού χωρί να γνωρίζει κανεί τον ιδιοκτήτη, ενώ ισχυρίζεται η εταιρεία ότι είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Κατά δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μεν εμπιστοσύνη, αλλά χρειάζεται χρειάζονται και ακριβείς πληροφορίες. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ως δεδομένο ότι αυτό που μας λένε οι εταιρείε για τους εαυτούς τους υπάρχουν αρχαία, υπάρχουν μητρώα που πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε αν οι εταιρείε, οι εν λόγω εταιρείε, είναι μικρομεσαίες. Στην έκθεση της Όλαφ αναφέρεται επίσης και ο έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, η οποία δεν εντόπισε ποτέ κανένα σφάλμα. Και το έχω πει και στο παρελθόν, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που διεξάγονται αυτοί οι έλεγχοι. Πρέπει να γίνουν ευφιέστεροι. όχι μόνο οριζόντιοι, αλλά και κάθετοι. Να εξετάζουν όλα τα αλληλοσυσχετιζόμενα στοιχεία. Συχνά πηγαίνουμε σε αποστολές ή επισκέψεις που μας λένε αυτοί που επισκεπτόμαστε ότι έχουν, λάβει, επισκέψεις, έχουν δεχτεί από 10 διαφορετικούς ελεγκτές και τελικά δεν έχουν εντοπίσει τίποτα οι ελεγκτές αυτοί. Η Όλαφ ε, δεν δήλωσε ότι υπήρξε απάτη και παρόλα αυτά η απάτη έγινε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι γιατί φοβόμαστε να δημοσιεύσουμε ε, το τελικό πόρισμα Ο Υπουργό Οικονομικών στην Τσεχία ή Υπουργό Οικονομικών στην Τσεχία είπε ότι θα συμβουλευτεί δικηγόρου για να ε, τη πούνε αν μπορεί να δημοσιεύσει την έκθεση ή όχι. Όμω δεν έγινε ποτέ καμία νομική πραγματογνώση για το θέμα. Εξ όσων γνωρίζω. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση θα μπορούσε και να δημοσιευθεί και να ενισχυθεί έτσι η εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δώσατε πολλά καλά παραδείγματα. Τα κονδύλια συνοχή έχουν βοηθήσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιε περιπτώσει όμω είναι ξεκάθαρα υποθέσει απάτη. Καλό θα ήταν κάποτε να συζητούσαμε και τι υποθέσει με θετική έκβαση και όχι μόνο τι αρνητικέ. Πάντω η γενική σα διεύθυνση μπορεί να αποφασίσει εάν οι Τσέχοι έχουν ε, ε, ολοκληρώσει έργα που ήταν επωφελή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Δημοκρατία της Τσεχίας. Ευχαριστούμε η συνάδελφος Λαμπάγιοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ω αντιπρόεδρο αυτή τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, ήθελα να σας ε, καλέσω να, παρακα... να παραμείνουμε πιστοί στις αρμοδιότητές μα που αρμόζουν στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο. Θέλω να σα θέσω τρει απλέ ερωτήσει, κύριε Γενική Διευθυντά, διότι είναι πολλέ οι λεπτομέρειε που αφορούν το έργο αυτό. Τρει ερωτήσει λοιπόν. Πρώτον, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το τελικό ποσό των δαπανών που δηλώθηκε δείχνει ότι το ποσό τη έρευνα τη Όλαφ δεν έχει σχέση με τη βοήθεια από το Ταμείο για την Ανάπτυξη, την Περιφερειακή Ανάπτυξη που θα πρέπει να πληρωθεί. Δεκέμβριο του 2018 θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό του. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι τσεχικές αρχές συμφώνησαν με τον ε, προτινόμενο υπολογισμό του τελικού ποσού με τις εκτόσεις του φετινού Ιανουαρίου, εάν δεν κάνω λάθος 25 τρέχοντος. Και τρίτη, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο φωλιά πελαργών και ότι δεν πρέπει να αναλυθεί καμία δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο δηλαδή. Κύριε Γενική Διευθυντά, γι' αυτό ακριβώς μας απασχολεί αυτό το θέμα, διότι αρχικά ε, ήταν ε, ένα ε, πρόγραμμα που για πολύ καιρό δεν είχε καταλήξει, δεν είχαν καταλήξει οι αρχές ότι έπρεπε να το βγάλουν από το πρόγραμμα στήριξη των επιχειρήσεων, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ήταν ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σημαντικό ε, για την Τσεχία και από πολιτική ε, πλευρά. και γι' αυτό μας, μας απασχολεί και εδώ και καιρό αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να δοθεί εντύπωση ότι μας αρέσει να τσακωνόμαστε με τους υπόλοιπους. Όχι, ήταν ένα πολιτικό ζήτημα. Μιλάμε εδώ για τις ε, βασικές αδυναμίες του συστήματος ελέγχου ε, στην ε, Τσεχία. Όταν ξεκινήσαμε το 2014 δεν υπήρχε καν απαγόρευση για συμμετοχή μελών της κυβέρνησης, που έχουμε πετύχει πολλά έκτοτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Τσεχία αλλά και για άλλες χώρες να έχουν πετύχει πλέον να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Κύριε Γενική Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Στεχόφσκι, νομίζω ότι μπορεί να είμαι πολύ σύντομος, δεδομένου ότι σας έχω ήδη δώσει πληροφορίες για το θέμα αυτό και στο, συζητώντας το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα ότι θα θέλαμε να έχουμε ε, αρκετές διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για μια μονομένη κατάσταση, η κατάσταση του Stork Nest. Και στο κλείσιμο της προηγούμενης περίοδου ζητήσαμε από τις ε, αρμόδιες αρχές να κάνουν ενδελεχή ελεγχό όλων αυτών των ε, σχεδίων τον ε, ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν στο παρελθόν δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο. Τώρα, επί του παρόντος, για την περίοδο 2014-2020. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που τα οποία είπατε. κάναμε μία κρόαση προληπτικά και σε αρχικό στάδιο για να εξετάσουμε, και αυτό είναι πέσει το Φεβρουάριο, όλες τις περιπτώσεις χορήγησης κονθυλίων που δίνονται στη Και είδαμε ότι η αρχή διαχείρισης καταρχάς ε, έδειχνε μεγάλη εμπιστοσύνη στις πρώτες προφορίες που έδειχναν οι διάφορες μιμίες. Τις περίφημες προφορίες πριν φάτσιε και έτσι δεν γινότανε συστηματική ενδελεχής ε, επισκόπηση του όλου θέματος μετά για τον καθένα, πράγμα το οποίο το κάνουμε τώρα. Και βεβαίως στα πλαίσια αυτή τη αλλαγή εκ μέρου μα είδαμε ποια ήταν η εξέλιξη άλλων προγραμμάτων τα οποία είχαμε ήδη υποστηρίξει. Δεν βρήκαμε όμως τέτοιου είδου περιπτώσεις εικονικών μημιέ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε το κατάλληλο σύστημα ελέγχων επιτόπου στην Τσεχία. Και το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις ε, αρχές διαχείρισης να ελέγχουν ε, τις ε, εταιρείες δικαιούχος. Όσον αφορά την δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Οι εκθέσεις της Όλαφ δεν είναι σαν όλες τις άλλες εκθέσεις και αναφορές. Και βεβαίως δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας. Κυρία Λαμπάγιοβα. Πρέπει να ομολογήσω δεν κατάλαβα το πρώτο ερώτημα που κάνατε. Το δεύτερο, ναι. Οι αρχές στην Τσεχία δέχθηκαν να αφαιρέσουν αυτό το πρόγραμμα από τα σχετικά προγράμματα της περιοχής τους. Και έκλεισε αυτή η υπόθεση. Προηγούμενο μήνα. Τρίτη ερώτηση. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι κοινοτικά κονδύλια δεν πήγανε στο Stock Nest die Entscheidung, die späte Entscheidung Ελήφθη καθυστερημένα η απόφαση και το θέμα είναι αν έχασε λεφτά η Τσεχία λόγω αυτής της κατάστασης. Ο απάντησε όχι. <clears throat> Δεν έχασε κάτι από το συνολικό ποσό της υποστήριξης με την απόσυρση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν πολύ καλή. Σας σας ξαναπροσκαλέσουμε. Πολύ καλά μας τα είπατε. Ευχαριστώ και την ομάδα σας ε, που ήταν εδώ όλη τη μέρα σήμερα και μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες και το λέω όχι ως απειλή αλλά ως ε, ανταμοιβή και ως ευχαρίστηση θέλουμε να σας ξαναδούμε. Θα μιλήσουμε σήμερα στις 2.30 ε, με τον κύριο Έτιγκερ για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν. Μέχρι τότε διακόπτουμε.